Θα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ανοίξει η διαδικασία των αιτιολογήσεων ψήφου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. πρώτη έκθεση είναι των, της κυρίας Παρβάνοβα και της κυρίας Χιμένεθ Μπεσερίλ Μπάριο με θέμα τα ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Ο κύριος Ρόντε έχει τον ε, λόγο. Κύριε Ρόντε, έχετε το λόγο. Med den øh, frie bevægelighed og den teknologiske udvikling, så er kriminaliteten i stadig højere grad blevet grænseoverskridende. Είναι θέμα, είναι γεγονός ότι η εγκληματικότητα τώρα έχει γίνει μια διασυνοριακή δραστηριότητα και ταυτόχρονα και οι διώξεις εις βάρος των εγκληματικών ομάδων γίνονται και αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν εγγύηση για τα δικαιώματα των θυμάτων οπουδήποτε στην Ευρώπη. Πρέπει να την χάνει κανείς προστασίας, φροντίδας, ε, διερμηνίας, μετάφρασης, νομικής βοήθειας κτλ. Εν μέρη υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση. Θα πρέπει να κινηθούμε όμως προς μια Ευρώπη πιο ασφαλή και μια ισχυρότερη αστυνομική συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Ήβα Ζανίκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ συχνά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θύματα μιας εγκληματικής ενέργειας δεν καταγγέλουν το γεγονός λόγω φόβου ή λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης. Στόχος του κειμένου είναι να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ε, θύματων της εγκληματικότητας να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε όλες τις χώρες της Ένωσης στρέφοντας την προσοχή μας στα θύματα τα οποία κινδυνεύουν να τύχουν περαιτέρω ε, ζημιών θα έλεγα ή βλαβών καλύτερα η αναγνώριση λοιπόν του καθαστώτος του θύματος όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι υπέστησαν κάτι μετά από μια παράνομη δραστηριότητα αλλά και για τους συγγενείς σαν παράδειγμα ενός θύματος που εξέπνευσε μετά ακριβώς την εγκληματική ενέργεια. Ε, δεν βλέπω την συνάδελφο κυρία Ματσόνη στην αίθουσα. Προχωρώ ε, στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Ρώση. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Τάσομαι υπέρ αυτής της έκθεσης ε, γιατί όταν μερικά χρόνια πριν ε, ήμουν ε, περιφερειακός σύμβουλος στο Πιεμόντε υπήρχε ένας νόμος για αναγνώριση αυτών που ήταν θύματα βίας και σε αυτή την περίπτωση αναφερόμασταν στο θα, ποιοι θα πρέπει να τύχουν προστασίας και κατά τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν κανονικά. Όλα τα θύματα θα πρέπει να την χάνουν να διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα και να την χάνουν της ίδιας προστασίας, να έχουν και τη δυνατότητα αποζημίωσης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα τα θύματα σεξουαλικής βίας και τους ε, ανήλικους σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, δίνω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υιοθετήσαμε την οδηγία για την υποστήριξη προς τα θέματα των εγκληματικών πράξεων. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χιμένας ε, τώρα οι γυναίκες οι οποίες πέφτουν θύματα βίας, διακίνησης ανθρώπων, θύματα τρομοκρατίας αλλά και κάθε εγκληματικής πράξης θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα του κράτους μέλους στο οποίο θα έχει διαπραχθεί αυτή η εγκληματική πράξη, ανεξαρτήτως της ε, πικότητάς τους. Θα έχουμε κοινέ λοιπόν προδιαγραφέ, σαφεί προδιαγραφέ που θα εξασφαλίζουν ε, τον χειρισμό με σεβασμό, αξιοπρέπεια και χωρί διακρίσει των θυμάτων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στην προσοχή που δίδεται σε παιδιά και σε άτομα με ειδικέ ανάγκε όπου θα γίνεται μάλιστα ιδιαίτερη αξιολόγηση του πόσο ευάλωτα μπορεί να είναι έτσι ώστε να μην ε, προξενηθεί, να μην δημιουργηθεί ε, μια ταξινόμηση των θυμάτων σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Πρέπει κύριε Πρόεδρε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό είναι ένα από τα δικαιώματα για τον κάθε πολίτη και με την οδηγία αυτή που αποτελεί ένα πρώτο καλό βήμα ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίησή της. Ο είναι συνάδελφος κύριος Μήτρο Ρέπο. Κύριος Μήτρο Ρέπο. Ε, Arvoisa puhemies, Ευχαριστώ πολύ. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, πολιτών είναι βασικό δικαίωμα των ε, Ευρωπαίων πολιτών και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κινούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκουν εργασία και να κινούνται ελεύθερα, να διακινούνται ελεύθερα. Πρόκειται για ένα βασικό και εκτιμένο και θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των πολιτών. Η μεταχείριση σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και η υποστήριξη καθώς και προστασία αν αποτελέσουν, ε, αν είναι θύματα βίας ή εγκλήματος γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ίση μεταχείριση και κοινή προστασία κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είμαι υπέρ των ε, βασικών δικαιωμάτων. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Βάντενχολτζερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πολιτική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτήν την εποχή αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα επιδείνωση των συνθήκων για πολλούς ε, πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία λοιπόν για τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας ε, θυμάτων εγκληματικών πράξεων δείχνει ότι οι αποφάσεις ε, δεν θα πρέπει πάντοτε να αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για εξέβρεση λύσεως. Επί παραδείγματι μια ομάδα θυμάτων, μια ομάδα ανθρώπων, τα θύματα αυτά δηλαδή, θα έχουν τη δυνατότητα για ισότιμη προστασία και ε, υποστήριξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως κράτους μέλους. Επίσης, ε, δημιουργούμε μια Ευρώπη της αντιμετώπισης των εγκληματικών πράξεων ανεξαρτήτως των προσωπικών δυνατοτήτων ε, των θυμάτων. Μια επαγγελματική δηλαδή βοήθεια χωρίς να γνωρίζει σύνορα, που δεν γνωρίζει σύνορα και που θα προσφέρεται στα θύματα αυτής της ε, εγκληματικότητα. Μια πολύ καλή μέρα λοιπόν για την Ευρώπη. Η επόμενη μιλήτρια είναι η συνάδελφο κυρία Κοστέλο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια φρικτή εμπειρία το να είναι κανείς θύμα ενός εγκλήματος. Η διαδικασία βέβαια της καταγγελίας και οι σχέσεις με τις αρχές εκ των υστέρων είναι και αυτό κάτι το πάρα πολύ δύσκολο μερικές φορές. Γι' αυτό λοιπόν η οδηγία αυτή, η οποία θέτει συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τους παρέχεται μετάφραση διευμηνία, Επίσης θα τους παρέχεται ανώνυμη και εμπιστευτική στήριξη σε όλα τα επίπεδα. Θα λαμβάνεται υπόψη επίσης το φύλλο τους, η εθνοτική τους καταβολή και γενικά ε, όλα τους τα επιμέρους χαρακτηριστικά. Θα βοηθήσουμε λοιπόν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύπτονται από τα δικαστικά συστήματα που διαφέρουν και υπάρχουν στα διάφορα σημεία της Ένωσης. Thank you. This report will ensure... Η έκθεση αυτή διασφαλίζει έτσι ώστε οι πολίτες οι οποίοι πέφτουν θύματα όταν ταξιδεύουν σε μια άλλη χώρα να τύχουν τις βοήθειες την οποία αξίζουν, την οποία χρειάζονται τους δίνει δυνατότητα πρόσβαση στην ενημέρωση και πρακτική υποστήριξη. Στο παρελθόν τα ξένα θύματα είχαν προβλήματα, είχαν εμπόδια στο να αποζημιωθούν ή να προστατευθούν πλήρως. Αυτά τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας τώρα θα καταστήσουν την κατάσταση πιο δίκαιη. Βασικές διαδικασίες με πιο συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Πρόκειται για μια καλή έκθεση γιατί πάρα πολλοί δυστυχώς θίγονται από τις καταστάσεις αυτές σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, Ο κύριο Τσάλ Τάνοκ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω πλήρω την θέσπιση ελάχιστων και ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την προστασία και υποστήριξη και τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πρόξεων. Παραδείγματι, το να λαμβάνει κανεί το αντίγραφο τη αστυνομική πράξη ε, στη γλώσσα που καταλαβαίνει ή να υπάρχει ενημέρωση και υποστήριξη προς τους οικείου των θυμάτων εγκληματικών πράξεων ή τρομοκρατικών ενεργειών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα οικογένειες να τοποθετούνται, να εκφράζονται στο δικαστήριο ακόμη και αν δεν είναι απευθεία μάρτυρες, εφόσον αυτό βέβαια δεν αντίκειται στις διαδικασίες. Ιδιαίτερα το πακέτο το σχετικό με τα δικαιώματα των παιδιών θα σημάνει μεγάλη πρόοδο προς την προστασία των παιδιών θυμάτων, ιδιαίτερα με τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω βίντεο συνδέσμου και όχι απευθεία μαρτυρία στο δικαστήριο. Είδαμε στην ε, ε, Γαλλία ένα αποτρόπαιο έγκλημα που άφησε ορφανά δύο παιδιά ε, βρετανική υπηκότητα, που πιστεύω θα αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία εφαρμογή αυτών των μέτρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα θύματα θα μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα επίπεδα δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να υπάρξει ένα συντονισμένο τρόπο αντιμετώπιση των θυμάτων. Πρόκειται για μια οδηγία τμήματο ενό ευρύτερου πακέτου, το οποίο θα βελτιώσει την ομοθεσία στον τομέα αυτό, έτσι ώστε τα θύματα των εγκληματικών ενεργειών να έχουν συγκεκριμένα πρακτικά δικαιώματα. Ε, ιδιαίτερα το πακέτο για την προστασία των παιδιών, το οποίο είχε προτείνει και ο κ. Σκέρκοπφ είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ε, Πάρα πολλά δικαιώματα λοιπόν των θυμάτων που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη οδηγία. Παρ' όλα αυτά θυμάμαι και νιώθω μάλλον απογοητευμένη ιδιαίτερα μετά από τις συζητήσεις που έγιναν σήμερα το πρωί που αναφέρθηκαν στο πόσο καλή είναι η Ευρώπη δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να επιβάλλουμε μια πανευρωπαϊκή ε, κατεύθυνση. Σαν ευρωπαϊκά κράτη αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να ανήκουν στους πολίτες μας χωρίς να είναι αυτό καταναγκαστικό. Νάρφος, κυρία Μακοβέη. Thank you, η πρόταση αυτή διότι θα ενισχύσει και θα δώσει περισσότερο περιεχόμενο στα περιεχόμενα στα, στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζουμε ελάχιστες προδιαγραφές για τα θύματα βίας και εγκλήματος ανεξάρτητα από την υπηκότητά τους ή από το που ε, έλαβε χώρα το έγκλημα. Θα πρέπει τα θύματα να έχουν τα ίδια δικαιώματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει η έννοια του θύματος, ο ορισμός να είναι ο ίδιος σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο κοινό ορισμός θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της δικαιοσύνης και θα υποστηρίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να υποστηρίξουμε τα θύματα εγκλήματος. Uh, θα δώσω τώρα το λόγο στον James Νίκολσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι η υιοθέτηση αυτή τη οδηγία είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την προσπάθεια την οποία έκαναν. Γνωρίζετε ότι προέρχομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία που έχουμε υποστεί δεκαετίες βίας από τους τρομοκράτες. Αυτό έχει επηρεάσει τις οικογένειες, ιδιαίτερα τις οικογένειες των θυμάτων αυτών των ενεργειών. Ελπίζουμε όλα αυτά να τα έχουμε αφήσει πίσω μας, αλλά δεν θα πρέπει να τα ξεχάσουμε και δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το πόσο έχουν επηρεαστεί οι ζωές τόσων ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι γιατί η έκθεση αυτή καλύπτει τις ανάγκες των θυμάτων της τρομοκρατίας, των οικογενειών τους και έχουν συγκεκριμένα πλέον δικαιώματα και υποστήριξη. Οι κυβερνήσεις έχουν δύο χρόνια για να μεταφέρουν την πρόταση αυτή στην νομική τους αρχιτεκτονική. Ζητώ το Ηνωμένο Βασίλειο να το κάνει το ταχύτερο δυνατόν γιατί επιτέλους η Ευρώπη όρισε σωστά το, το, την έννοια του θύματος, κάτι το οποίο ε, θα βοηθήσει πολλούς από τους κατοίκους της χώρας μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο ρόλος και οι ανάγκες των θυμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη επαρκώς από την Εθνική Ένωμη Τάξη. Πολλές φορές ε, τα θύματα δεν την χάνουν σωστής και αξιοπρεπούς μεταχείρισης και γι' αυτό δεν μπορούν να έχουν σωστή πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δικαίωμα αποζημίωσης. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της υποστήριξης θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος χαρακτήρας και αμοιβαία αναγνώριση από όλα τα κράτη-μέλη. Άρα οι δικαιοδοτικές αρχές αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συστή σωστή και ενιαία υποστήριξη των θυμάτων. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτή την έκθεση και θεωρώ ότι με την έγκριση αυτής της οδηγίας θα βελτιωθεί η κατάσταση των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα την χάνουν των ίδιων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Δίνω συνάδελφο Ντάνιελ Χάναν. Κύριε Πρόεδρε, ένας κλέφτης που δρά αυτόνομα είναι απλώς ένας εγκληματίας. Αλλά μια συμμορία κλεφτών προσπαθεί να ελέγξει την ε, ε, οικονομία των χωρών ε, μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά. Ο ληστή λοιπόν ο μεμονωμένο, μπορεί να πάει φυλακή. Αλλά οι τραπεζίτες, η οργανωμένη αυτή ε, συμμορία ληστών συνεχίζει ανενόχλητη να κλέβει τα χρήματα των πολιτών. Και μας λένε μετά οι υπουργοί μας ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα χρήματά μας σε αυτούς τους συμμορίτες, σε αυτούς τους ληστές και να ε, περιμένουμε πότε θα έρθει η ώρα της ταξιοδότησης. Έχουμε πια ξεφύγει από την ε, αρχή της ευημερία, έχουμε ξεχάσει την αρχή της ευημερία και επικρατεί παντού η φτώχεια στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα με την Νομισματική Ένωση. Στα 20 χρόνια που εορτάζουμε φέτος από την έξοδο της χώρας μου από την Νομισματική Ένωση μπορούμε... Πάλι εκτός θέματος. Πάλι είστε εκτός θέματος κύριε Χάναν. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο συνάδελφο κύριο Καμάλ. Thank you very much, Mr. Vice President. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Νομίζω ότι αυτά, αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που ενώνει το σώμα μας όλοι τασόμαστε υπέρ των θυμάτων, ιδιαίτερα όταν τα μέτρα δεν είναι επαρκή και όπου βλέπουμε ότι τα θύματα δεν έχουν τα δικαιώματα με τους ε, ημεδαπούς ενός κράτους μέλους. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είναι εύκολη η εναρμόνιση για κάτι επί του οποίου συμφωνούμε. Λέμε ας εναρμονίσουμε διότι μας ενδιαφέρει η τύχη των θυμάτων, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ανήλικα. Θα πρέπει όμως να μην είναι η αρχή ενός ολισθήματος υπέρ της εναρμόνισης των δικαιωμάτων. Καταρχήν πιστεύουμε σε αυτό το δρόμο, αλλά όταν γίνεται ολιστηρό το έδαφος, πού κινούμαστε ως προς τα δικαιώματα των κρατών μελών. Ε, επόμενο θέμα ε, είναι η έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ, μέτρα κατά των χωρών, οι οποίες επιτρέπουν την διεξαγωγή μη βιώσιμης με στόχο τη διατήρηση των ηχθιαποθεμάτων. Αιτιολογής ψήφου, δίνω μέσα το λόγο στον ε, συνάδελφο κύριο Σαλβατόρη Γιακολίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα έγιναν δεκτές, ε, αν όχι συγκεκριμένες προτάσεις ή τουλάχιστον η επιθυμία διαβεβαιώθηκε πλέον του Κοινοβουλίου για να υποστηρίξει την αντιαυτική δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Εγώ υπερψήφισα την πρόταση αυτή γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο μέσω της περιφερικοποίησης να υπολογιστούν με τον καλύτερο τρόπο οι δυνατότητες παρέμβασής μας. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τη δραστηριότητα αυτή, να αυξήσουμε τις διεξόδους διάθεσης των προϊόντων και να διασφαλίσουμε θα έλεγα μια συγκεκριμένη σύγχρονη ανάπτυξη ενός τομέα ο οποίος ε, συνδυάζει την περιβαλλοντική αηφορία με την οικονομική παραγωγικότητα. Και γι' αυτό θα πρέπει μέσω των ταμείων που ελέγχουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να επιταχυνθεί η βελτιωτική αυτή διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω τις χώρες οι οποίες ε, δεν αλλιεύονται, δεν αλλιεύουν συγγνώμη με τρόπους που καταστρέφουν το περιβάλλον σύμφωνα και με τις απόψεις ε, του κόμματός μου σε σχέση με την ε, αηφόρο παραγωγή ε, προϊόντων και την διάθεση των τροφίμων. Έχουμε προβλήματα σε σχέση με την υπερβολική αλίευση σκόμβρων σαν παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καλύψει όλα τα αλλιεύματα τα οποία ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο θα έλεγα αλλιευτικό περιβάλλον και σχετικά με την επιβολή αυτών των περιορισμών και δράσεων εγώ είμαι υπέρ της προσπάθειας αξιολόγησης των κοινωνικών συνεπειών των μέτρων αυτών έτσι ώστε τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται λοιπόν να είναι δίκαια και να είναι και συμβατά με τις υποχρεώσεις της Ένωσης απέναντι στον ΠΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά μια εποχή όπου να κοινή αλληλευτική πολιτική και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα και τι δραστηριότητε των αλλήλων μα, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί και ισότιμη αντιμετώπιση προ τι εισαγωγέ των αλληλευμάτων. Και εγώ υποστήριξα την πρόταση αυτή ε, γιατί επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις ε, εισαγωγές από, προϊό, από περιοχές ε, όπου δεν γίνεται βιώσιμη αλίευση από τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω γιατί με τόσο ενθουσιασμό υποστήριξα την πρόταση. Διότι υπήρξε η εποχή όπου ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταγράψει τη βόλωση του Κοινοβουλίου. Αποτέλεσε δηλαδή μια ισχυρή ψήφο του Κοινοβουλίου, μια ισχυρή τοποθέτηση και πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου και πρέπει η Επιτροπή να βρει τρόπο να καταστήσει τις θέσεις μας συμβατές και με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και όχι να μας λέει το αντίστροφο ότι λόγω των ε, διεθνών υποχρεώσεων δεν μπορεί να τηρηθεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Next speaker is ε, Mr. Ο κύριος Higgins είναι επόμενος ομιλητής. Υποστηρίζω στεναρά αυτή την έκθεση. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για να έχουμε πραγματικά βιώσιμες αλλιευτικές πρακτικές που αφορούν τα αλλιευτικά αποθέματα και τη σωστή τους ε, χρήση. Θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις σε κράτη που οδηγούν στην υπερεκμετάλλευση αλλιευτικών αποθεμάτων ή που δεν συνεργάζονται σωστά μέσα στα πλαίσια των συμπεφωνημένων. Εμείς έχουμε αναφέρει κατά κόρο ότι θα πρέπει να αποστείλουμε ένα δυνατό μήνυμα προς την Κομισιόν ότι δεν θα δεχτούμε συναλλαγές με χώρες που δεν προβάλλουν τη βιώσιμη αλία, διότι εμείς μόνο θα χάσουμε η δική μας αλία και τα ε, δικά μας αλλιευτικά προϊόντα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη μη βιώσιμη αλία και τα προϊόντα θα πρέπει να απαγορευτούν τα σχετικά προϊόντα. Ναι, Ο κύριος Γιάρ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και βεβαίως εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ λογικό να θέλει κανείς να επιτρέπει την αλία μόνο όριμων ε, ψαριών. Δυστυχώς όμως πολλές φορές ο άνθρωπος δεν ορθολογικά και γι' αυτό πρέπει να παρεμβαίνουμε και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της υπεραλίευσης, γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τους αλίες μας και στις παγκόσμιες, σε, σε όλες τις θάλασσες και επίσης θα πρέπει να ε, αντιδρούμε απέναντι σε εκείνου, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν σέβονται αυτές τι βασικές αρχές της λογικής αλλίευση. Γι' αυτό λοιπόν ε, συμφωνώ και εγώ με την πρόταση, ευχαριστώ του συναδέλφου που την υπερψήφισαν και πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και να επισημάνει στα κράτη αυτά τα οποία προβαίνουν σε υπεραλίευση ότι είναι πολύ σημαντική η βιώσιμη αλίευση, γιατί δεν αφορά μόνο εμάς, δεν αφορά μόνο τους αλίες μα, αλλά πάνω απ' όλα το μέλλον και τις επόμενες γενναίε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάννη. Είναι η συνάδελφο κυρία Έλενα Μπασέσκου. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece eforturile Uniunii Europene de a realiza activități de pescuit sustenabil nu sunt suficiente cât timp sunt singulare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 Επί της εκθέσεως του συναδέλφου κ. Στίβερσον με θέμα κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Καλώς το βήμα τον κύριο Τσάρλ Στάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, θα ε, ήθελα να πω ότι εγώ υπερψήφισα σε σχέση με την οργάνωση των αγορών, την ε, κοινή οργάνωση αγορών, την έκθεση του κυρίου Στίβενσον, που πιστεύω θα πρέπει να προστατεύει τους, ε, τις οργανώσεις των καταναλωτών και επίσης θέλω να αναφερθώ στον στόχο των οργανώσεων καταναλωτών με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασία ιδιαίτερα στι περιοχέ τη Υπέθρου, αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση που θα δώσει κίνητρα στου νεαρού ε, ε να μπουν στο επάγγελμα. Πρέπει να δοθεί λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αλίας και θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ε, ανάγκη να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί ο πολίτης και ενδεχομένως να δημιουργηθεί και μία, και μία ε, ευρωπαϊκή ετικέτα προϊόντων. Ο κύριος Μέρφυ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ στήριξε την πρόταση αυτή. Η κοινή οργάνωση αγορά θεσπίστηκε τη δεκαετία του 70 με στόχο να εξασφαλιστεί ένα καλό δίκαιο εισόδημα για τους αλληλείς. Δεν εξασφαλίστηκε όμως ποτέ αυτός ο στόχος. Καταψηφίζω λοιπόν και την έκταση Χάγκλοντ για την εκμετάλλευση των λευτικών πόρων. Ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα καταστρέψει τους σπόρους. Οι μικρές και μεσές αλληλευτικές μονάδες θα κατακριστούν από την, ε, τους μεγάλους αλληλευτικούς στόλους που θα απορροφούν όλο το αλίευμα. Πρέπει πιστεύω να ξαναθέσουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της αλίας και της διαχείρισης των αλληλευτικών αποθεμάτων και πρέπει να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα για τους αλίες μας και βιώσιμη διαχείριση αυτών πόρων. Αυτή η έκθεση είναι η πρώτη από τρει νομοθετικέ προτάσει τη Κομισιόν για την μεταρρύθμιση τη κοινή ελευτική πολιτική και θέλει να δώσει κίνητρα στην αγορά για να υποστηρίξει τι βιώσιμε πρακτικέ και να ενισχύσει το δυναμικό τη αγορά των ε, ευρωπαϊκών προϊόντων. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε πιο βιώσιμη αλία βέβαια, αλλά επίσης πρέπει να υποστηρίξουμε τους αλείς παράλληλα. Ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών δεν μπορεί να υποτιμηθεί σε αυτή την εξίσωση. Και καλωσορίζω την εισαγωγή σαφών στόχων, ούτως ώστε να προωθούν επικερδείς και να απορρίψουν την ασίδωτη αλία. Επίσης, θα πρέπει να μην υπάρχουν παραλιεύματα και θα πρέπει να υπάρχει να γίνεται η άσκηση αλληλεία με έναν υπεύθυνο τρόπο χωρί να στραβλώνεται η αγορά. Επίση, υποστήριζω ε, ε, του συναδέλφου και τι τροπολογίε, του κύριου Στίβενσον, ούτω ώστε να υπάρχει μια οικολογική ετικέτα για τι βιώσιμε πρακτικέ στην αλληλεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω όλα αυτά λοιπόν και ελπίζω να καταφέρουμε ότι η νέα κοινή αλληλευτική πολιτική ε, πετυχαίνει αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Jim Higgins. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγή τον κύριο Στίβενσον για μια πάρα πολύ, έκθεση, πάρα πολύ καλή έκθεση με πολύ διάλογο, τροπολογίες και συμφωνία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για τον ρόλο των οργανώσεων καταναλωτών στα άρθρα 6, 2, 32 και επίσης στις κοινές προδιαγραφές στα άρθρα 32 και 34. Όσον αφορά την ε, σταθεροποίηση της αγοράς, η Κομισιόν επιτέλους αναγνωρίζει την τεράστια διακύμανση των τιμών στον τομέα. Έχουμε τώρα επιτέλους έναν κατάλογο ε, ψαριών που μπορούν να καταψυχθούν, ε, να γίνουν παστά και να αποθηκευτούν με διάφορους άλλους τρόπους. Ε, οι ελάχιστες αυτές προδιαγραφές σημαίνουν πως οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν επιλογές με βάση τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 42-46. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν ένα κλειδί για την επιλογή του τέλος. Καλωσορίζω τις διατάξεις του άρθρου 49 που χρειάζονται για να αντιληφθούμε καλύτερα την αλυσίδα αυτή της παραγωγής και της τάσης αγοράς. Ε, επόμενη είναι η κυρία Έλενα Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση γιατί θα πρέπει νομίζω να εξασφαλίσουμε υψηλό βαθμό προβλεψιμότητα στι οργανώσει παραγωγών. Η κοινή οργάνωση αγορά, του τομεί των προϊόντων αλληλεία αντιπροσωπεύει μια συνιστόσα πολύ σημαντική τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Η επιλογή των προϊόντων που πρέπει να γίνεται με τα λόγου γνώσεως είναι πολύ σημαντική για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Η χρήση μιας ε, βιολογικής ε, ετικέτας για τα αλληλευτικά προϊόντα δίνει τη δυνατότητα σαφών πληροφοριών σε ό,τι αφορά την, το βιολογικό χαρακτήρα και την ημερομηνία λήξη των προϊόντων. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει συνάφεια μεταξύ της κοινή πολιτικής του τομέα της αλίας και της κοινή εμπορικής πολιτικής τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην ενωσιακή αγορά θα πρέπει να σέβονται τα ίδια πρότυπα εμπορίας και θα, με αυτά που σέβονται δηλαδή οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Η επόμενη έκθεση είναι του συναδέλφου κυρίου Μπροκ με θέμα ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Στάνοκ εξ ονόματος της ομάδας ECR. Σας ευχαριστώ. Η ομάδα μας αποδέχεται την πραγματικότητα της ε, ΚΕΠΑ και την ανάγκη βεβαίως να μπλεκούμε σε αυτήν, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει ανάγκη της ομοφωνίας στο Συμβούλιο, καθώς δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπονομεύσει την εθνική κυριαρχία, η οποία θα πρέπει να παραμείνει στα Εθνικά Υπουργεία Εξωτερικών. Γι' αυτό απήχε η ομάδα μου. Και όσον αφορά όλες τις πτυχές της έκθεσης Μπροκ. Βεβαίως ε, είδαμε επικοδομητικά τις, ε, ε, τα αιτήματα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και με μάτι κριτικό, ειδικά όσον αφορά τα μη ρεαλιστικά αιτήματα αύξησης του υπερπολογισμού σε αυτούς τους καιρούς λιτότητας. Και βεβαίως πρέπει να γνωρίσουν πως η υπηρεσία λειτουργεί. Αλλά στο κλίμα αυτό της λιτότητας πρέπει να αποδείξει την προσθέμενη αξία της και με εξοικονομήσεις των μικρότερων κρατών μελών και να και σε μεγάλα κράτη όπως το δικό μου το Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία θα πρέπει να δουν πώς το εθνικό του συμφέρον προστατεύεται και προβάλλεται καλύτερα μέσω της νέας υπηρεσίας. Ένα καλό παράδειγμα είναι το νέο ευρωπαϊκό συγκρότημα στο Νέο Σουδάν όπου θα εγκατασταθούν σε μια κοινή πρεσβεία όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης αναφέρθηκε και η Ταϊβάν και η δέσμευσή της για την ειρήνη και τη συνεργασία και την ασφάλεια στην περιοχή. Επίσης ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πρωτοβουλία του Προέδρου της ε, χώρας αυτής ε, για την νότια Συνική θάλασσα και δύο συγκροτήματα νησιών. Οι εντάσεις πρόσφατα κλιμακώθηκαν καθώς χτες νομίζω η Κίνα απέστειλε ακτεωρούς σε αντίδραση κάποιων κινήσεων της Ιαπωνικής κυβέρνησης. Το φιλόδοξο σχέδιο του Προέδρου της ε, Ταϊβάν, κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τη συνθήκη της Ανταρκτικής, νομίζω πως αξίζει τη στήριξη. Το λόγο έχει συνάδελφος κυρία ε, Νόρικα Νικολάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Είναι μια ετήσια έκθεση. Είναι μια έκθεση ένα έντυπο θέσης, είναι ένα έγγραφο το οποίο θα πρέπει να παρουσιάζει ένα όραμα. Συνεχίζει στην κλασική όμως άγουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να υπάρχουν πολλές καινοτομίε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να βλέπω ότι για τη συνιστόσα της ασφάλειας της ευρωπαϊκής πολιτικής ο εισηγητής μίλησε για σημαντικά θέματα, έθιξε σημαντικά θέματα, όχι μόνο για το μέλλον της κοινή πολιτικής, αλλά και για την ε, σημασία, για την ορατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τα σύνορά της. Εδώ μιλάω για την ενίσχυση του δυναμικού της υπηρεσίας αυτής εξωτερικής δράσης που δρά και για την πρόληψη των συγκρούσεων. Νομίζω ότι το να υπάρχει ένα αντίστοιχο προπολογισμό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, θα ήθελα να μιλήσω για το εμπόριο όπλων στα πλαίσια των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την μελλοντική μας επιτυχία. Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα αυτή την έκθεση και θα ήθελα να αιτιολογήσω το γιατί. Πρώτα απ' όλα να μην ξεχνάμε πως ε, υπάρχει η άποψη των ε, συναδέλφων ε, που μιλάνε για μια στρατιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής και μια ε, σύμπλευση με τον ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο για μένα ως Αυστριακό δεν είναι αποδεκτό. Αλλά πρέπει να δούμε και την ε, κατάσταση με την ε, Τουρκία και απαιτείται εκεί πέρα το να ανοίξουμε περαιτέρω ε, κεφάλαια στη διαπραγματευτό ότι απέτυχε η υπόθεση τη ε, Λιβύη. νομίζω είναι πλέον ξεκάθαρα, έχει αποτύχει τελείω η πολιτική εκεί πέρα, είδαμε και τι έγινε στην ε, Βενγάζη και η πολιτική μα στη Συρία επίση απέτυχε, είναι μια πολιτική η οποία στρέφεται κατά της Ρωσίας, της Κίνας, εταίρων μας δηλαδή και όλα αυτά γιατί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα θέλουν να αναλάβουν την εξουσία στην Συρία. Μα οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε την ε, διάλεκτο της Σαουδικής Αραβίας. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κ. Σέρτζιο Γκαετάνο Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Έρμαρ Μπρόκ αλλά παρόλα αυτά δεν αποκρύπτω τις μεγάλες δυσκολίες και τα όρια της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να τονίσω δύο στοιχεία τα οποία με ανησυχούν όλος ιδιωτέρως. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το εμπόριο όπλων. Ε, θέλουμε, έχουμε θέσει το στόχο του μη πολλοπλασιασμού, τον αφοπλισμό και παράλληλα έχουμε διατάξεις που είναι εντελώς ανεπαρκείς ό,τι αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων. Επομένως, αυτό που λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε το αρνούμαστε, το ακυρώνουμε με τη συμπεριφορά μας και με τις διατάξεις μας. Δεύτερο θέμα, ε, όπου φαίνονται τα όρια μας με τρόπο καταφανή είναι ε, η πρόληψη των συγκρούσεων που θα πρέπει να μας επιτρέπουν να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Αυτό που συνέβη στην ειρήνη. Αυτό που ονομάσαμε ακατάλληλα και λανθασμένα αραβική άνοιξη. Εμείς καθυστερήσαμε ως συνήθως. Δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε σε αυτέ τι χώρε. Δεν ήμασταν σε θέση με την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγουμε να φτάσουμε σε καταστάσει δραματικέ ό,τι αφορά α, τη ζωή των ανθρώπων. Ελπίζω στο μέλλον η εξωτερική μα πολιτική να είναι πιο αποτελεσματική σε ό,τι σε, ό,τι, σε σχέση με τα, αυτό που ήταν τους τελευταίους μήνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοφεράτη. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Γιάννους Ζέμκε. Ε, bardzo chciałem podziękować. Ε, po przyjęciu traktatu w Lizbonie... Ε, Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την ε, υιοθέτηση της συνθήκης Λισαβόνας ε, υποτίθεται πως θα ενίσχυε την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία. Η πρόοδος είναι πάρα πολύ αργή. Καλές είναι οι προθέσεις, αλλά τα γεγονότα ελάχιστα. Αυτό μπορεί να εκφραστεί από την δραστηριότητα διαφόρων ομάδων ε, στην Ευρώπη διαχείριση δε αυτών των ομάδων μάχης των λεγόμενων ευρωπαϊκών υπάρχει μόνο στα χαρτιά και επιχειρησιακά δεν έχει γίνει τίποτα. Ε, οπότε δεν ε, υπάρχει ακόμα πεδίο στρατιωτικής ε, συνεργασίας. Πρέπει λοιπόν να προγραμματίζουμε από κοινού σε μεγαλύτερη κλίμακα και να κάνουμε αποστολές και στρατιωτικές επιχειρήσεις από κοινού. Πρέπει να συνδυάζουμε την ε, στρατιωτική δράση με τη συνεργασία στην στρατιωτική βιομηχανία και θα ενθάρρυνα εδώ πέρα την Κομισιό να αναλάβει πιο φασιστικά βήματα. Ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Άνταμ Μπίλαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ απήχα σε αυτή την ψηφοφορία αυτής της έκθεσης για διάφορους λόγους. Μιλάμε για την άμεση χρήση πόρων, για αυτή την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Φυσικά θέλουμε να, υπάρχει, να υποστρίξουμε τη σχέση μας με τη Μόσχα και φυσικά είμαστε υπέρ της ε, σημασίας της στρατηγικής σχέσης με τη Ρωσία. Επίσης είναι πολύ σημαντική η σχέση μας με την Ταϊβάν, αλλά οι προτάσεις της έκθεσης να αυξήσουμε το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μας προβληματίζει. Υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή μας μέσω της εξωτερικής υπηρεσίας ε, αυτής. Δεν μπορούσα λοιπόν να συμφωνήσω 100% με όλη την έκθεση. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κ. Γιάνν Κοσλόφσκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για κατά την άποψή μου. Είναι ένα στρατηγικό και φιλόδοξο έγγραφο. Θεωρώ πως ε, καθώς η πολιτική γειτονία είναι κύριος στόχος της πολιτικής ασφαλής ένωσης ε, ήταν σωστή αυτή η κίνηση. Είμαι ικανοποιημένος ε, από αυτά τα οποία αναφέρονται για την συνεργασία με τις χώρες ανατολικής γειτονίας και παρά τις ανησυχητικές δραστηριότητες στην νότια γειτονιά μας θα υπάρξει κάποια ισορροπία και η ανατολική διάσταση θα συνεχίσει να μας απασχολήσει. Να μας απασχολεί. Τέλος, η έκκληση στην ύπατη εκπρόσωπο να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις αποστολές παρακολούθησης ε, των εκλογών στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Ευχαριστώ. Πολύ ε, Το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοί μου, υποστήριξα και εγώ την έκθεση του Έλμαρ Μπρόκ. Ε, εμείς μέχρι τη συνθήκες αποκτούμε νέες εξουσίες, αλλά υπάρχουν νέες εξελίξεις, νέες κρίσεις, νέα γεγονότα, ε, τη υπόψη και της οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά σημαίνουν μια μείωση του ενδιαφέροντος που έχουμε για την γειτονία μας. Το σχάρι η στα κράτη της Αραβικής Άνοιξης. Αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος συγκεκριμένα συντάσσει ένα νέο σύνταγμα. Δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με αυτά τα τεκτενόμενα. Έχουμε νέες εκλογές στη Γεωργία. Υπάρχουν παγωμένες συγκρούσεις, όπως το Αμπόρνο Καραμπάχ και αλλού. Υπάρχει μια κάποια κόπωση θα έλεγα με την κατάσταση της Ουκρανίας. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να αποστρέψει το, τα μάτια του από την πολιτική γειτονία. Δίνω το λόγο στην άδελφο κυρία Έλενα Μπασέσκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα την έκθεση του κυρίου Μπροκ γιατί βεβαίως η επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων μπορεί να γίνει μόνο με τρόπο συνολικό. Η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια σειρά μέσα που τις επιτρέπουν να μιλάει με μια φωνή αλλά εξακολουθούμε να έχουμε αρκετές ελλείψεις όσον αφορά την ΚΕΠΑ. Η εδραίωση σχέσεων μεταξύ της ε, ε, υπηρεσίες εξωτερικής δράσης Κομισιών και των κρατών μελών ακόμα δεν υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνεργασία όσον αφορά δε το μέλλον της ε, ΚΕΠΑ πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ανατολική διάσταση. Η ανατολική αυτή εταιρική σχέση θα πρέπει να προωθήσει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς Ανατολάς ε, και σε νέες χώρες όπως η Μολδαβία. Είναι του συναδέλφου κ. Χάγκλουντ με θέμα διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων. Αιτιολογής ψήφου. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Τσάλ Στάνοκ. Από το 2002 η Κομισιόν ήταν υποχρεωμένη με βάση κανονισμό του Συμβουλίου να λογοδοτεί για τους αλληλευτικούς πόρους και για τους περιορισμούς ε, που υπάρχουν και αυτό πρέπει να το κάνουμε μέχρι το 2011. Ε, η έκθεση λέει ότι υπάρχουν προσπάθειες από τα κράτη-μέλη για να διατηρήσουμε τους πόρους μας, αλλά δεν είναι επαρκείς αυτές οι προσπάθειες και λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για τη μείωση του αλληλευτικού δυναμικού. Είμαι υπέρ της έκθεσης γιατί λέει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει, υπάρξει συγκεκριμένο ορισμό του αλληλευτικού δυναμικού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ε, θα πρέπει να έχουμε ορισμού για τα περιφερειακά θέματα και μηχανισμού συλλογή δεδομένων, ε, καθώ και μακρο, μακρόπνοα σχέδια, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν με αυστηρότητα. Έχουμε ένα τριπλό νομοθετικό πακέτο, το οποίο όμως δεν καταφέρει να πετύχει αυτά που πρέπει. Ε, τότε θα πρέπει να αμφισβητήσουμε όλη την κοινή αλλιευτική πολιτική και να την επανεθνικοποιήσουμε. Είναι η τελευταία απόπειρα για να διορθώσουμε τα πράγματα για τους Ευρωπαίους αλληλείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση παρά το ότι πάντα είμαι επιφυλακτικός όταν ακούω τη λέξη διατήρηση. Σκεφτόμαστε δηλαδή το περιβάλλον χωρίς τις ανάγκες των αλλιέων. Η έκθεση αυτή όμως είναι διαφορετική. Είναι σαφές πως ε, τα κρατη θέλουν να ενισχύσουν την διατήρηση και να ε, ενισχύσουν τα αλλιεύματα κάτι το οποίο δεν είχαν κάνει μέχρι στιγμής παρά τη μείωση των αλευτικών στόλων. Το σύστημα των ε, περιορισμών στα ύδατα, στα 12 ναυτικά μίλια λειτουργούσε αρκετά καλά και νομίζω μπορεί να επεκταθεί και στα 20 μίλια για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ε, πρέπει οι ψαράδες να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το γιατί υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί καθώς πάρα πολύ συχνά ο αυτοπεριορισμός είναι η μοναδική ρεαλιστική λύση. Αλλιώς δεν θα αντιμετωπίσουμε την υπεραλίευση. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις ενώσεις ε, των αλλιέων και τα περιφερειακά ληφτικά συμβούλια και όλους τους ενδιαφερόμενους για να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα προστασίας του οικοσυστήματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο στηρίζω. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία, η κυρία Έλληνα Μπασέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση γιατί το σημερινό σύστημα των αλληλευτικών ποσοστώσεων ε, κατέδειξε τα προβλήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Η βιωσιμότητα του αλληλευτικού τομέα έγινε δευτερεύον θέμα. Για να επιλύσουμε και να διορθώσουμε τα προβλήματα θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να περιφερειοποιήσουμε την αλληλευτική πολιτική ούτω ώστε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκινήσει ε, μακροπρόθεσμα προγράμματα που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών και παράλληλα να λάβουμε υπόψη μα την ανάγκη να διατηρηθούν ε, οι αληθικοί πόλοι. Ε, πάνω από 60% των αληθικών πόλων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεραλλιεύονται πάνω από το μέγιστο όριο αντοχής. Ε, αυτό επηρεάζει και άλλα είδη όπως τα δελφίνια στην Μαύρη Θάλασσα τα οποία ε, ψαρεύονται κατά λάθο στα δίχτυα. Έχω κάνει λοιπόν μια γραπτή δήλωση για την ανάγκη να προβλέψουμε μέτρα προστασίας των δελφινιών στη Μαύρη Θάλασσα. Αδέλφω αυτή του συναδέλφου κύριου Νικολάου Σαλαβράκου με θέμα μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ο κύριος Αντρέα Ζανώνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής είναι μια αναγκαία επιλογή. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Συχνά ε, ψαρεύουμε πολύ και άσχημα. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τους ε, βιολογικούς θαλάσσιους πόρους, να διατηρήσουμε το θαλάσσιο σύστημα και να εξασφαλίσουμε την ε, βιωσιμότητα του κλάδου, θα πρέπει να σταματήσουμε την υπεραλίευση διαφόρων ειδών. Ε, επίσης, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να, κρατήσει το, να διατηρηθεί το, κράτο, το status quo ε, και παραλίγο να περάσει αυτό. Εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη μεταρρύθμιση, μια συνεπή μεταρρύθμιση που επιτρέπει μια βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων ε, και παράλληλα πρέπει να έχουμε και προοπτικές για το μέλλον. Πρέπει να έχουμε ε, πολυετή ε, προγράμματα και θα πρέπει να έχουμε δίκτυα προστατευόμενα Επίσης θα πρέπει να έχουμε κυρώσει για τα κράτη-μέλη τα οποία δεν σέβονται τους κανόνες, που δεν ελέγχουν, που δεν σέβονται τις ποσοστό του και που δεν είναι αξιόπιστα στοιχεία. Μεγαλύτερη ε, προστασία ε, σημαίνει περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τους ε, αλίες μας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα που δεν το έχουν καταλάβει. Ο κύριος, κύριος Uh, uh, uh, η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής σημαίνει τώρα πως η Κομισιόν θα ενθαρρυνθεί με τρόπο μη δεσμευτικό να ενισχύσει μέτρα διατήρησης των αλληλευτικών πόρων, κάτι το οποίο συμφωνεί με την στρατηγική του κόμματός μας για την βιοπικιλότητα και ελπίζουμε να υπάρξει και οικονομική βιωσιμότητα, κάτι το οποίο συμφωνεί με το υπεύθυνο οικονομικό μοντέλο που προτείνουμε εμείς για να υπάρχουν δουλειές στον τομέα αυτών και τέλος να προωθήσει την περιφερειακή πολιτική, κάτι το οποίο συμφωνεί και με τον εθνικό μας στόχο στο Ηνωμένο Βασίλειο για διαμοιρασμό των ευκαιριών μεταξύ περιφερειών. Η κοινή αλληλευτική πολιτική, όπως είπα, κατά την άποψή μου, είτε θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να εξυγχρονιστεί δραστικά, είτε να εγκαταληφθεί εντελώ από τις αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το λόγο έχει ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ικανοποιημένο που αυτό το σχέδιο ψηφίσματο υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να έχουμε μια συνεπή και στραφή στρατηγική για το μέλλον, ούτως ώστε οι αλείς να προγραμματίζουν τις επενδύσεις μέσα σε κλίμα ασφάλειας. Ο τομέας υδατοκαλλιέργειας, αν τον διαχειριζόμαστε σωστά, με βιώσιμο τρόπο θα μπορούσε, όπως λέει το ψήφισμα, να συνεισφέρει περισσότερο στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας, να εξασφαλίσει ασφάλεια τροφίμων, ποιότητα, απασχόληση, προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση ε, μιας δυναμικής αλληλείας, ε, καθώς και των παράκτιων ε, κοινοτήτων. Είμαι Ιρλανδός και είμαι πολύ ικανοποιημένο που το ψήφισμα λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να διερευνήσει την ε, μείωση του, της αλίευσης των αλλιευτικών πόρων και θα πρέπει να έχει ε, προγράμματα διαχείρισης ούτως ώστε να βλέπουμε την κατάσταση των αλλιευμάτων ε, και αυτό αποκινούμε τα εμπλεκόμενα και ενδιαφέρομενα κράτη-μέλη. Η συνάδελφος κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Η μεταρρύθμιση της αλίας στην Ευρώπη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικότητες στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια σειρά από μελέτες και έρευνες για να δούμε τα διαθέσιμα αλληλεύματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε εκτιμήσεις για τη βιώσιμη αλληλεία, και βιώσιμο τρόπο αλληλείας αυτών των αλληλευμάτων. Οι εκτιμήσεις θα πρέπει να προβλέπουν και χρονοδιαγράμματα, τόσο ώστε να μειώσουμε την αλληλεία, την αλληλευτική προσπάθεια δηλαδή, με σκοπό την ανανέωση των αλληλευτικών πόρων σε ένα βραχυπρόθεσμο διάστημα. Είναι σημαντικό αυτές οι μελέτες να προσαρμόζονται ε, στις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους και να λαμβάνουν υπόψη ε, το πραγματικό αλληλευτικό δυναμικό. Η δυνατότητα περιφερειοποίησης της αλληλευτικής πολιτικής επίσης θα πρέπει να αναλυθεί πιο προσεκτικά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε ότι τα αλληλευτικά κονδύλια χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπασέσκου. Ε, δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Chris Davis. E Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε από τα μέλη του ΕΛ και τα αλλού Ιρλανδού Ισπανού Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ξέρουν τι κάναμε σήμερα. Ξέρουμε πώ εξαλούνται τα ε, αποθέματα, αλλά σήμερα ψήφισαν τροπολογία που λέει πω δεν θα ε, βοηθήσουμε να ανακάμψουν τα αλλιεύματά μας. Να το ξαναπώ. Υπερψηφίσαμε τροπολογία του ΕΛΚ που λέει πως δεν θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να ανακάμψουν τα αλλιεύματα. Ε, φαντάζομαι ότι το έκαναν για τους καλούς ε, λόγους που θέλουν να δοθεί άλλος ένας χρόνος στον κλάδο. Αλλά ο μόνος τρόπος βεβαίως να γίνει αυτό είναι να δώσουμε λίγο χρόνο στα ψάρια, στα αλλιεύματα. Μόνο έτσι έχει μέλλον η αλλία. Δεν ξέρω τι θα σκεφτούν οι πολίτες μας. Θα σκεφτούν πως αυτή η πτέρυγα εκεί πέρα είναι παλαβή, παλαβή άνθρωποι. Είστε τελείως τρελοί. Έχετε δύο μήνες να το ξανασκεφτείτε μέχρι να ψηφίσουμε οριστικά αυτή την νομοθεσία. Ε, τελευταία, τελευταία ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση δίνει μια επισκόπηση της θέση του Κοινοβουλίου ε, στην πρόταση της Κομισιόν για μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής. Τα μέτρα για την συντήρηση, τη διατήρηση των πόρων ε, με βρίσκουν σύμφωνοι. Αλλά αυτή η έκθεση μα δείχνει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια επιχειρήματα θα ακουστούν του επόμενου μήνε. Είδαμε, ήταν μια πρώτη γεύση. Θα υπάρξουν επιχειρήματα και συμβιβασμού για τι λέξει. Υπάρχει μια τροπολογία για μια απόπειρα να αλλάξουμε κάποια πράγματα πάνω από την μέγιστη απόδοση, ε, κοντά στη μέγιστη απόδοση. Επίσης, ε, μιλάμε για την ανανέωση, αλλά στην πραγματικότητα θέλουμε να δώσουμε δημόσιο χρήμα για να αντικαταστήσουμε ε, σκάφη, να τα κάνουμε μεγαλύτερα, με υψηλότερο δυναμικό και όχι κατά ανάγκη να φτιάξουμε πλοία τα οποία βοηθούν στην διατήρηση των λευτικών πόρων. Ε, θέλω να δουλέψουμε πάνω στη μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσει αυτή τη βιωσιμότητα. Ε, χάρη όμως τις τροπολογίες που πέρασαν, εγώ δεν μπόρεσα να υποστηρίξω αυτήν την έκθεση. Κύριε κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση διακόπτεται. Επανέρεξη της συνεδρίασης σε 35 περίπου λεπτά. Ευχαριστώ.